σε σχέση με τις στάση της Επιτροπής ΕΚΟΝ για την ε, έκφραση διαδικασίας αντιρρήσεων σε ό,τι αφορά εφαρμοστικές εκτελεστικές πράξεις που έγιναν πριν από την έναρξη της παρούσας ε, ολομέλειας, δεν υποβλήθησαν ε, αντιδράσεις μέσα στην 24ωρη προθεσμία. Με βάση το άρθρο 105 ε, παράγραφος 6 του εσωτερικού κανονισμού, οι συστάσεις της ΕΚΟΝ ε, θεωρούνται εγκεκριμένες και θα δημοσιευθούν στο κείμενο των πρακτικών της σημερινής ε, ημέρας, δηλαδή από την Τετάρτη